θα κάνουμε ένα, ένα τεστ να λειτουργεί. Λοιπόν, έχουμε μυστική ψηφοφορία, δοκιμάζουμε. Όποιος θέλει μπορεί να πατήσει όποιο κουμπί θέλει. Δηλαδή, να δει αν λειτουργεί το σύστημα. Μόνο τεστ είναι αυτό, δεν κάνουμε τίποτα. Λειτουργούνε. Ωραία. Satu is from Helsinki, where Escher has the seat, so you have... Σάτου είναι από το Ελσίνκι, έχει, έχει, εκεί την έδρα τη. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα, ε, έχουμε δύο υποψήφιους. Από ό,τι κατάλαβα, το ναι σημαίνει μία από τις υποψηφίους και το όχι την άλλη. Και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι τι. Σας παρακαλώ μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Για ποιον θα ψηφίζουμε με το ναι και με, σε ποιον όχι. Και εγώ είμαι ε, το άτομο επαφής με την υπηρεσία αυτή της ΕΧΑ για, τα χημικά, για τις χημικές ουσίες. Θα ήθελα να σας πω ότι εκείνος που θα εκλεγεί σήμερα ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο θα δράσει κυρίως ε, σε επαφή και ενημέρωση της ε, Επιτροπής. Γιατί οι εκπρόσωποι που είχαμε μέχρι στιγμή δεν έκανε τη δουλειά του τόσο καλά. Ωραία, ευχαριστώ αυτό. So you spoke in favor of Christine. Λοιπόν, εσείς εκφραστήκατε υπέρ της Χριστίνα Ρουντέν. For για την κυρία Λεπερούς, μήπως θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, ο Κρίς. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται να είμαι υπέρ κάποιου και δεν νομίζω ότι έκανε και κάτι αντίστοιχο η αλλά συμφωνώ απόλυτα με την άποψή τους ότι οποιοδήποτε διοριστεί θα πρέπει να επικοινωνεί με την Επιτροπή πολύ περισσότερο από τον προκάτοχό του. Εξαιρετικά. Α, ωραία. Τώρα κατάλαβα πώς θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε και όποιο έχει την πλειοψηφία θα είναι η μα. Τώρα ακούστε με προσεκτικά. Κριστίνα Ρούντεν ρο θα έχουμε red root. Λοιπόν, Οποιο θέλει να υπερψηφίσει την Κριστίνα Ρούντεν θα πρέπει να, ε, να πάρει το κόκκινο κουμπί. Το κόκκινο. Όποιος θέλει να υπερψηφίσει για την Άννα Περούς, το πράσινο παρακαλώ. Αριστερά δηλαδή. So we have one vote. Λοιπόν, διαμιά θα ψηφίσουμε. Όποιο θέλει να ψηφίσει υπέρ τη Κριστίνα Ρούτεν θα ψηφίσουμε στο δεξί μέρος, εκεί που είναι το κόκκινο και όποιοι θέλουν να υπερψηφίσουν την Άντλα Περούς, το πράσινο που είναι στο αριστερά. Με συγχωρείτε. Είμαστε πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά είναι πολύ περίπλοκο για τα μέλη που έχουν εξαντληθεί στη διάρκεια της χρονιάς. Αριστερά για τη Λαπερούς λοιπόν και δεξιά για τη Ρούντεν. Ορίστε. It's not green or red. Λοιπόν, όχι green or red, left, right. Left, Λαπερούς, right, Ρούντεν. Μυστική ψηφοφορία λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποια σύγχυση, διότι στον κατάλογο ψηφοφοριών με αλφαβητικά σειρά έχουμε τους δύο υποψήφους. Εσείς αρχίζετε από το δεύτερο στη σειρά, το αναφέρω στους συναδέλφους για να μην κάνουν λάθος ψηφίζοντας, διότι συνήθως ψηφίζουμε τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά. Δεν είναι ο Ρούντεν που πρέπει να ψηφιστεί πρώτος. Νομίζω ότι είναι σαφή. τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, right και left. Μία ψηφοφορία και για τους δύο υποψηφίους μυστική ψηφοφορία. left. left <laughs>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 35 ψήφους για την κυρία Λεπερούς και 23 ψήφους για την Κριστία Ρούντεν και μία αποχή συνολικά. Λοιπόν, ορίζουμε την κυρία Λεπερούς να μας εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑ στο Ελσίνχη, της Υπηρεσίας της Χημικής Ουσίας. Και θα της δείσουμε να επικοινωνεί το στενότερο δυνατό με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ωραία. Η εύκολη ψηφοφορία ήταν αυτή. C'était clair. Ah, Περνάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 20. Ενεργειακή απόδοση. Έχουμε τον εισηγητή μας Πίτερ Λίζε εδώ. Oh so, we start with the vote. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, λέει ο κ. Λίζε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου οι οποίοι βοήθησαν επίση τη γραμματεία και του συνεργάτε που μα βοήθησαν. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του Σκιώδη είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γραμματότηση γιατί ζητήσετε τη μελλοντική μα πολιτική για το κλίμα. Ήταν δύσκολο να πετύχουμε συμβιβασμού, τελικά όμω έτυχαν ευρεία υποστήριξη. Έχω μία παράκληση μόνο. Μετά από πολλέ και μακρέ συζητήσει, έχουμε ένα συμβιβασμό για το 19 και την ελληνική σκέψη 34 για το σύστημα εμπορίου εκπομπών, του ETS και προτείνουμε μία πολύ μικρή παρέμβαση. Είναι, όπως σας λέω, ένας πολύ επιφυλακτικός ε, τρόπος ε, παρουσίασης. Και αν ψηφίζαμε ξεχωριστά και την τροπολογία 353 θα ήταν αντίθετη με, ε, με το πνεύμα γιατί θα έβαλε και και στις ε, επιχειρήσει οι οποίε τηρούν τι τις ε, Εάν δεν πετύχουμε λοιπόν το συμβιβασμό που θα ήθελα να σα παρακαλέσω να το υπερψηφίσουμε, θα ήθελα να καταψηφιστεί η 354. Δηλαδή θα πρέπει να καταπέσει ή θα πρέπει να καταψηφίσουμε η 354. Πρώτος, ωραία, είχε διευκρινιστεί αυτό. Είχαμε την εντύπωση ότι είναι ξεχωριστά η τροπολογία αυτή. Τώρα ακούσαμε τι είπε ο από αυτού. Ο καθένα θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσει κατά συνείδηση. Ευχαριστώ Πέτερ για το σχόλιο σου. Περνάμε στην πληροφορία τώρα. Τροπολογία 18. Ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επτά. υπέρ με την προφορική τροπολογία ναι ενοποιημένη επτά με προφορική τροπολογία υπέρ η προφορική τροπολογία θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά δεν είναι τμήμα του συμβασμού πρόεδρε α εντάξει ο συγητής είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Κοιτάξτε. Είναι αντίθετο με τον συμβασμό, γι' αυτό είμαι κατά. Α, ωραία. Καταπίπτει άρα. Θα ψηφίσουμε τώρα την ενοποιημένη τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πενιδευτά Σαμπίνα Βίλς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 απεσύρθη. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 70 Ευχαριστώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται, να. Και περνάμε στην. Πέντε. Άρθρο 3α νέο. Τροπολογία 5 του εισηγητή. Υπέρ. Τροπολογία 5. 3α νέο άρθρο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε. Άρθρο 5 παράγραφος 1. Τροπολογία 135. Ζήπε. Υπέρ. Ένα λεπτό. Για να προσανατολιστούν όλοι στο κείμενο. 135. Τροπολογία 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Παρακαλώ. 136 σκυλακάκης θέλει να ελέγξει γιατί δεν είχε πλειοψηφία. Ελέγχουμε την 136. Und beendet. Πέρας ψηφοφορίας. Σχεδόν, παραλίγο. Δεν άρχισε όμως. 134. 134. Παναγιώτοφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το άρθρο 6 παράγραφο 5 σημείο Γ τροπολογία 162 Βλάχο των Μποντορόφ Παναγιώτοφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Άρθρο 11 παράγραφος 1. 296 Ορέστε Ρώση και 297 Γιάννο Σάνταρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 299 υπέρ. Τα κατά αποχές απορρίπτεται 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές ελέγξουμε Δεκτομικός έλεγχος Alle abgestimmt, beendet. τη ψηφοφορία. Α, υπέρ, υπέρ, ναι, εγκρίθηκε. 315, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 316, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 317, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 318, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 321 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 fällt weg. 325 καταπίπτει. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Und die Μία ψήφο φιλελευθέρω δεν αρκεί να αλλάξει την πλειοψηφία. Λοιπόν, 333 υπέρ. Και 334 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την 354, τη γνωστή. Θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ 354. Κατά. Να το ελέγξουμε αυτό. Abstimmung beendet. Πέρας. 30 προς 28 με μία αποχή εγκρίνεται. Wir kommen zu den Annexen. Παραρτήματα τώρα. 360 υπέρ. Κατά. Συγχωρείτε, δεν πρόσεξα να ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. 460. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 363 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...364 με 367. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 368. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 369. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 370. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 374. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 376. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 378, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 381 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 385 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 387 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 390. Ελέγχουμε 390. Abstimmung beendet. Πέρασε Ναι, απερίφθη. Πράγματι. 391. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 393-394. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 395 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 396 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 398 υπέρ κατά αποχές Απολύπτεται. 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 401 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 403 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 405 υπέρ απεσύρθη η άλλη απεσύρθη στην οποία αναφέρεστε 405 έχουμε φτάσει υπέρ της 405 κατά να ελέγξουμε Τη 405. Beendet. Πέρας. Απερίφθη. 406. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 407. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 407. Und beendet. Abgelehnt. 408. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 410. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 411. Υπέρ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 αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την 37 να ελέγξουμε την 37 Beendet. Ναι, ναι. Απερίφθη πράγματι η 37. Συγγνώμη. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. όχι, 42, συγγνώμη, 42 Κρήτον Αρσένης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα, μπορούμε ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε πάνω στο σύνολο της τροποποιημένης πρότασης. Άρχεται ψηφοφορία. Abstimmung beendet. Πέρασε τη ψηφοφορία. 52 υπέρ, 3 ε, κατά, 6 αποχέ. Συγχαρητήρια, Πέτερ Λίζε. Yeah. Arbeit... Για την τόσο ουσιαστική εργασία και ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την προετοιμασία τη ψηφοφορία. Yeah, ein wichtiger Bericht. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Το επίκεντρο της Δανικής Προεδρίας στο επόμενο εξάμεινο θα είναι. Ja, wir machen weiter mit. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για δικού ιατρικού σκοπού. Hallo, Peter. Peter Liese. Hallo.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 Λοιπόν, ελπίζω η συζήτηση για την ενεργειακή απόδοση μπορεί να συνεχίσει εκτός της αίθουσας, παρακαλώ. Are you all ready for the next point? Είσαστε έτοιμοι για το επόμενο σημείο? Και ο, ήδη, και ο και ο Θεόδρος Κυρακάκης ξέρουν τι κάναμε μέχρι τώρα. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα στη μερική διάταξη. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συγγήτρια να μας κάνει μια παρουσίαση, η Φρεντερίκε για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ας αρχίσουμε. Ε, σήμερα είναι κάπως γιορταστική η ατμόσφαιρα. Είναι η μέρα αυτού του κανονισμού, εφόσον όχι μόνο συζητείται εδώ για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και οι δύο επιτροπές για γνωμοδότηση. Σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούν από το θέμα ο κ. Σταπουλά στην Ήτρε και η συνάδελφο Ινβάνοβα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Αρχίζω λέγοντας ότι θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω, θα μιλήσω εδώ για τα ουσιαστικά σημεία. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το 77, λεπτά Δεν πρόκειται να σας μιλήσω για 30 χρόνια ιστορίας. Για πάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε προβλέψει τις μεγάλες διατροφικές τάσεις που άρχισαν να διαφαίνονται με την εμφάνιση των πρώτων διαιτητικών τροφίμων προσπάθησε να νομοθετήσει για αυτά τα προϊόντα τα οποία ονομάζονται διαιτητικά και με την πάροδο του χρόνου αυτή η νομοθεσία συμπληρώθηκε και τώρα υπάρχουν 7 κείμενα τα οποία διέπουν αυτό το θέμα. Τα περισσότερα κείμενα υιοθετήθηκαν σε επιτροπολογία και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ε, όλες τις λεπτομέρειες. Δεν θα σας την οδηγία 4 για τα τρόφιμα, για μια ειδική ε, διατροφή υποθερμιδική για την ανοχή στη γλουτένη, για τις ε, ουσίες, ε, τις προσθετικές για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς, η ετοιμασία για νεογνά προϊόντων που εξάγονται κατόπιν, επίσης για τα νεογνά και τα προϊόντα, τα υγρά και τα προϊόντα τα στέρεα. Εδώ, 30 χρόνια αργότερα, είναι η ώρα των λογαριασμών για την Επιτροπή και για μας και αν πιστέψουμε τις 66 σελίδες του Impact Assessment που είναι πάρα πολύ διαφωτιστική αξιολόγηση, οι λογαριασμοί αυτοί δεν είναι συνολικά ικανοποιητικοί. Δύο απόψεις δακτυλοδεικτούνται πρώτα απ' όλα ο κατατεμαχισμός της εσωτερικής αγοράς, ένας διπλωματικός τρόπος για μένα για να πω ότι ορισμένες επιχειρήσεις κάνουν νομοθετικό shopping δηλαδή. Εποφελούνται πράγμα που είναι νόμιμο σήμερα από την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στην νομοθεσία για τα διατητικά προϊόντα με ε, το, την, το κανονισμό Herflains ε, του 2006 για τις βιταμίνες ε, και ε, το άλλο για τα συμπληρώματα διατροφής. Κάτι άλλο επίσης στην έκθεση που, ε, που κατηγορείται είναι η λιγότερη αξία για τον καταναλωτή του οποίου η αγορά ε, ε, δικαιολογείται από μια ειδική ανάγκη να χάσει βάρος, ανοχή ή όχι σε ορισμένα σε ουσίες. Τι δικαιολογεί αυτή την αγορά και το να πληρώσει ακριβότερα ένα διαιτητικό προϊόν που απλώ ενισχύεται με βιταμίνες ή με άλατα, μεταλλικά άλατα, ενώ ε, δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό από ένα κανονικό τρόφιμα. Συμπέρασμα για την Κομισιό είναι ότι αυτή η αντίληψη του διατητικού προϊόντος δεν έχει λόγο ύπαρξης και προτείνει να κατηργηθεί αυτός ο ορισμός, αυτή η φιλοσοφία και θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτή την βούληση καλύτερης νομοθεσίας ε, νοικοκυριού κατά κάποιο τρόπο αυτή η βούληση εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων που λήφθηκαν ο κανονισμός πάνω στον οποίο εργαστήκαμε πολύ για την ε, σήμανση Food ε, Information for Consumer ή τους επόμενους κανονισμούς για το 2012 που θα κωδιδοκοποιήσει ορισμένους ισχυρισμούς υγείας, δηλώσεις υγείας ε, μετά την ε, Επιτροπή της Διατροφικής Αλυσίδας. Η Επιτροπή προτείνει σε αυτήν την βούληση διευκρίνησης και απλούστευσης εφεξήσα τα διαιτητικά τρόφιμα να εξαρτώνται από το, και τον κανονισμό 2006 για τις ε, δηλώσεις που μπορεί να είναι κάπως ριζική αυτή η δήλωση και διατηρεί ένα, με τρεις τύπους για τα νεογνά και τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, υγρά και στερεά και τα τρόφιμα ε, για τους ε, ε, ασθενείς που βρίσκονται κάτω από ιατρική επιτήρηση. Οι πληθυσμοί λοιπόν, οι ευπαθείς, οι ευάλωτοι θα ωφεληθούν από αυτούς τους ειδικού κανόνες που αναφέρονται στη σύνθεση και στην ετικετοθεσία, στη σήμανση των διαφορετικών αυτών τροφίμων σχετικά με τους ισχυρισμούς με τις δηλώσεις στις τροπολογίες 23 και 46 προβλέπονται μόνο για, τις, ε, ε, για τα σκευάσματα για τα βρέφη. Με τους σκιώδεις εισηγητές εργαστήκαμε ε, για τα έγγραφα αυτά, συνήντησα τον κύριο Σίτερ για τους πράσινους, την κυρία Ντολόν για την Ελκ Ζαρμπό, για τους σοσιαλιστές Γιώτα, για την Κούε και την κυρία Γκίλινγκς ε, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Είχαμε μαζί μια ανταλλαγή καρποφόρος ε, και θέλω να εντάξω στο κείμενο μερικές από τις ανησυχίες τους. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι ουσιαστικό για μας να έχουμε όλες αυτές τις προοπτικές και να ενισχύσουμε τις διατάξεις που υπάρχουν ε, και που αφορούν ε, τις ε, πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Αυτή η νομοθεσία και το τονίζω γίνεται τηρώντας την αρχή της προφύλαξης, τροπολογίες 13, 14 κλπ. και πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην τυχαία παρουσία παρασιτοκτόνων Μιλάμε εδώ για βρέφη και για άτομα ε, υπό ειδική ιατρική επιτήρηση. Έχουμε κατόφλια όρια και έχουμε και την εκπροθέσεως παρουσία που πρέπει αυστηρά να απαγορεύεται στροπολογίες 43-45 όπου τήρησα όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το γράμμα των υφισταμένων νομοθεσιών στον τομέα αυτό νομίζω ότι οι πολίτες θα σοκάροντο εάν η νομοθεσία ευρωπαϊκή επιτρέπει παρασιτοκτόνα σε προϊόντα για τα οποία μιλάμε για την ώρα, δηλαδή για τα βρέφη. Δεν είναι μόνο ε, τα παρασιτοκτόνα, αλλά και τοξικές ουσίες και άλλες οικογένειες χημικών προϊόντων, διοξίνες Υπάρχουν και άλλες χημικές ουσίες και είναι σημαντικό να τις επισημάνουμε, να τις αναφέρουμε και να τις αποκλείσουμε. Τρίτο σημείο, η κυρία Ζάργο και η κυρία Λιωτάρ επέμειναν ότι είναι σημαντικό και ο κύριος Περιγιώ δεν είναι πλέον εδώ διότι μόλις τελειώσαμε την ομοθεσία για τους χυμούς πορτοκαλιού ήταν μια μάχη σε διάλογο τριμερές ε, ή να έχουμε ίδιους κανόνες, ίσους όρους για τα προϊόντα που εξάγονται και εισάγονται. Αυτό φαίνεται προφανές αλλά καμιά φορά και τα προφανή πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Τροπολογία 35 και 42 τέταρτο και αυτό ε, δεν αφορά μόνο την ομάδα των φιλελευθέρων. Σκεφτήκαμε τις πιο δυναμικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αυτές που αποτελούν ε, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, την καρδιά, τον πυρήνα του τομέα και αυτές που συνήντησα δεν είναι πολύ ικανοποιημένες με την πρόταση όπως έχει τώρα. Δηλαδή τα προϊόντα αυτά να περάσουν στην νομοθεσία Health Claims ε, θελήσαμε να ακούσουμε τις ανησυχίες τους. Δεν πρόκειται μόνο για ασφάλεια τροφίμων και για υγεία, αλλά και για κόστος. Είναι σημαντικό να μιλάμε για κόστος για μια μικρομεσαία επιχειρήση, να γίνει δεκτή από την ΕΦΞΑ μια, ένας ισχυρισμός, μια δήλωση ε, είναι ένας κόστος μεταξύ των 500.000 και του 1 εκατομμυρίου ευρώ για να γίνει δεκτή, δεκτός ένας ισχυρισμός, μια δήλωση. Όλες αυτές οι ε, σκέψεις με έκαναν να προτείνω τρεις ουσιαστικές αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τις ειδικέ διατάξεις σχετικά με την υποθερμιδική ε, δίαιτα. Είναι ένας ε, τομέας καινοτόμος. Ακόμα πιο σημαντικό προτίθεμε να προτείνω της very low calorie, ε, δηλαδή τα προϊόντα με πολύ χαμηλές θερμίδες, ε, τις περιλαμβάνω στον ορισμό των προϊόντων για γιατρικούς σκοπούς. Δεν χρειάζεται να έχουμε ασάφεια για τους πληθυσμούς που τρέφονται μόνο με αυτά τα προϊόντα. Ο ορισμός περιλαμβάνει τα προϊόντα από 400 έως 800 θερμίδες. Είναι πληθυσμοί που είναι βάλωτοι όταν παίρνουν μόνο αυτά τα προϊόντα Έλαβα ε, μια παρατήρηση από το λόμπι, ακούω όλες τις γνωμοδοτήσεις και καταλαβαίνω πολύ καλά ότι έχουν σημασία. Αλλά όταν ακούω να λέγεται ε, στα επιχειρήματα ότι εδώ ε, στιγματίζουμε με αυτά τα μέτρα ε, τους παχύσαρκους, τους όλο και περισσότερους παχύσαρκους που αυξάνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο και ότι η παχύσαρκία δεν είναι ασθένεια. Το 2001 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, την ανέφερε ως ασθένεια και εμείς το κάναμε το 2008. Αυτό για να σας πω ότι ορισμένα επιχειρήματα είναι αμφισβητήσιμα. Τρίτο σημείο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Ναι, ναι, κλείνω, κλείνω, κλείνω θα πρέπει τα τρόφιμα που είναι για όλα τα άτομα που πάσχουν από ε, έλλειψη ανοχής για τη γλουτένη. Ε, έχουμε επίσης ε, για την λακτόζη και για άλλα θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο νομικό που να είναι σταθερό και αυτό είναι και το, το, οι παρατηρήσεις του Συμβουλίου. Η νέα ε, νομοθεσία Somers για την σήμανση των Food Information for Consumers που στο άρθρο 36 προέβλεπε να, ε, να τονιστεί η σημασία ε, της συμπερίληψης αλλεργιογόνων στα προϊόντα και αυτό αφορά τη γλουτένη και την λακτόζη. Αυτά για να κλείσω η αναγκαιότητα να προβλέψουμε το πιο ασφαλές νομικό πλαίσιο με συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για τους ευάλωτους και στοχοθετημένους πληθυσμούς. Δεν χρειάζεται να ξαναγράψουμε τον νόμο, αλλά να εφαρμόζουμε καλύτερα τα υφιστάμενα κείμενα ως προς την πρόσβαση το, του κοινού στα επίσημα έγγραφα και την διαφάνεια που είναι κάτι σημαντικό για τον κύριο Σλούτερ και ε, σχετικά με την γενική ε, νομοθεσία περί τροφίμων που βασίζεται στις αρχές διαφάνειας και προφύλαξης. Έκλεισα, το κάνω στην, ε, σε αιτιολογικές ε, σκέψεις ευχαριστώντας ε, τα όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και ε, στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, ε, η Γραμματεία, Σκιώδη, Σκιώδης, συγητές που ανέφερα, όλα τα μέλη των λόμπι, όλους τους ενδιαφερόμενους, τους εμπλικόμενους, τους νομικούς γλωσσολόγους του Κοινοβουλίου που μελέτησαν τις τροπολογίες και θα ήθελα την βοηθό μου Πατρίσο Ντιβέρ να την ευχαριστήσω που έχει ένα μωρό τριών ετών και ένα μωρό που θα γεννηθεί λοιπόν ε, θα ενδιαφέρεται η ίδια για τα τρόφιμα ε, που προορίζονται για τα βρέφη. Θα ακούσω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια σας. Αρχίζω με τους σκιώδεις συγητές. Να σα επισημάνω ότι έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη, επομένω πρέπει να είμαστε σύντομοι. Τρία λεπτά για του σκιώδει, η Έστεν Λάγκεν η πρώτη. Τρία λεπτά μου φτάνουν. Τέσσερι παρατηρήσει. Καταρχά, νομίζω ότι η γενικότερη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να προσπαθήσει να εξορθολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι μια καλή προσέγγιση. Νομίζω ότι ο έλεγχο ο οποίο πρέπει να γίνει από πλευρά μα είναι ε, ποιε ομάδε ανθρώπων είναι τόσο ευάλωτε ώστε να δικαιολογείται να υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη σύνθεση των τροφίμων που καταναλώνουν. Νομίζω ότι για τα βρέφη είναι σαφέ αυτό. Είναι επίσης σαφέ όταν πρόκειται για ιατρικούς λόγους και θα πρέπει να υπάρξει και η συζήτηση για τις δίαιτες πολύ χαμηλές ε, σε θερμίδες για το κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτέ σε αυτό το πλαίσιο. Ε, γίνεται επίση μεγάλη συζήτηση για τρόφιμα τα οποία βρίσκονται στα κράτη-μέλη σε αυτό το πλαίσιο και θα βρεθούν εκτός βάσει αυτής της διαδικασίας εξορθολογισμού. Κατά την άποψή μου, ο βασικός έλεγχος ε, είναι να μην αλλάξει τίποτα για τον καταναλωτή. Δηλαδή, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνε που εφαρμόζονται για τη χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένι, για παράδειγμα, θα παραμείνουν οι ίδιοι, ώστε να μπορεί να είναι κάποιο βέβαιο ότι είναι ίδια η σύνθεση του τροφίμου που καταναλύνει, ανεξάρτητα από το αν ε, βρίσκεται σε ένα ε, ειδικό σύστημα ή στο γενικότερη νομοθεσία για τα τρίφωμα, ε, τρόφιμα. Πέραν αυτού, βέβαια, δεν μπορούμε να επιλύσουμε το σύστημα των αποζημιώσεων μέσω των ασφαλιστικών ασφαλιστικών συστημάτων στα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία απόπειρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό για τα ε, γάλατα διατροφής, το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, τα βρεφικά γάλατα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα τρόφιμα θα βρίσκονται εκτός ε, της ε, βασικής νομοθεσίας, που για μένα είναι καλή προσέγγιση, αλλά τι θα αλλάξει για τον καταναλωτή. Εγώ δεν θέλω να απαγορεύσω αυτά τα προϊόντα. Εάν κάποιος θέλει να πληρώνει ε, μεγάλα ποσά χρημάτων για ένα προϊόν ενώ Κάποιοι άλλοι μπορεί να πούνε ότι τα παιδιά άνω του ενό έτου μπορούν να πίνουν κάλλιστα το ίδιο γάλα, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δυσανεξία, ε, τότε έχει καλώ. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Τι θα γίνει όμω αν αυτά τα προϊόντα δεν ανήκουν πλέον σε αυτή την νομοθεσία, θα μπορούν να ε, καλύπτονται από τη γενικότερη νομοθεσία για τα τρόφιμα ή θα αλλάξουν τα πράγματα για τον καταναλωτή. Η ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίση ε, τι γίνεται με την ε, ε τρέχουσα κατάσταση. Τα γάλατα τα οποία επιτρέπονται αυτή τη ε, στιγμή στην αγορά είναι τα ίδια. Υπάρχουν διαφορές για τα κράτη-μέλη. Κάποια εντάσσονται στη μία κατηγορία και κάποια στην υπόλοιπη ε, νομοθεσία. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα ε, συνεχίσει η διάθεση των προϊόντων αυτών, αλλά κατά την άποψή μου εκτός του εξειδικευμένου κανονισμού. Τελό κάτι εξίσου σημαντικό, επειδή ακριβώς ο τομέα είναι πολύ επιστημονικός, ε, τα θέματα καινοτομία ε, ε, μπορεί να πρέπει να ληφθούν υπόψη και να πρέπει να δεχτούμε και τα νέα τρόφιμα στην αγορά. Και μία ερώτηση και πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τι έχουμε ρυθμίσει ήδη και τι χρειαζόμαστε όσον αφορά την επιπρόσθετη προστασία. Εγώ δεν θα ήθελα να ξαναρχίσει η συζήτηση για την φυτοπροστασία και τη σχετική νομοθεσία εδώ. Το να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασία για τα βρέφη και τους ασθενείς, ε, ναι μεν, αλλά δεν θα ήθελα να ξαναγίνει η ίδια συζήτηση για την φυτοπροστασία και τα προϊόντα αυτά. Τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή στον τομέα αυτό. Η Λίντα Μακάβαν, η οποία αντικαθιστά το σκιώδη εισηγητή, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν μπορεί να είναι η σκιώδη εισηγήτρια. Μου έδωσε κάποιε σημειώσει, αλλά επειδή δεν είμαι ειδική επί του ζητήματο, αλλά άκουσα πολύ προσεκτικά την εισηγήτρια, θα ήθελα απλώ να πω ότι όπως και η συγγήτρια χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνούμε για τη γενικότερη κατεύθυνση, για τα πιο συγκεκριμένα τώρα θέματα. Για τα βρεχηφικά τρόφιμα θέλουμε δράση για τα ε, φυτοφάρμακα, ιδίω για τις βρεφικές τροφές. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα... Δεν ξέρω γιατί ακούγεται αυτός ο θόρυβος, δεν έχει κανείς... Ε, θα αλλάξω μικρόφωνο, λέει ο μιλήτρια. Um, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, να μπορεί να μας εξηγήσει γιατί θέλουν να αλλάξουν οι κανόνες εισαγωγής ε, και εξαγωγής προς τρίτε χώρες. Θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές για τη σύνθεση που έχουμε ε, και με τα δικά μας προϊόντα ζητά επέκταση σε θέματα διαφήμισης, τα οποία ισχύουν για τις βρεφικές τροφές, να ισχύουν και για τα ε, υπόλοιπα στοιχεία, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους γονείς. Υπάρχει πολλές φορές έμεση διαφήμιση. Να σας πω ότι εγώ πήγα να πάρω ε, βρεφικό γάλα για την ανιψιά μου και διαπίστωσα ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει έμεση διαφήμιση στα ε, προϊόντα για μωρά άνω των 6 μηνών. Υπάρχει επιφύλαξη τώρα για τα προϊόντα αυτά, το τι θα πρέπει να ρυθμίζεται με τα διαιτητικά προϊόντα τώρα, τι πρέπει να εμπίπτει σε αυτό τον κανονισμό και τι πρέπει να εμπίπτει στους ισχυρισμούς για τα τρόφιμα. Ε, τώρα, τρόφιμα για ειδικού ε, ιατρικούς σκοπούς, ε, η σκιώδη εισηγήτρια θέλει να παραμείνει αυτή η κατηγορία και υποστηρίζει τις υπολογίες της εισηγήτριας να είμαστε ε, σε ένα στενό πεδίο εφαρμογής και να διαβεβαιωθούμε ε, ότι τα πάντα καθορίζονται βάσει των ισχυρισμών τροφίμων. Θα πρέπει να υπάρχουν και ε, κατάλληλες πληροφορίες ε, για το ιατρικό προσωπικό και τους επαγγελματίες, αλλά θα πρέπει αυτές οι πληροφορίες να παραμένουν για αυτούς και όχι να περνούν τους καταναλωτές. Τώρα, οι ΜΕΣ ε, θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για να μπορούν κατόπιν να συμβουλεύουν γονείς και ασθενείς. Τα διατητικά τρόφιμα, κατά την άποψη της κοιόδησης ηγήτριας, δεν ε, απαιτούν ειδική κατηγορία, ε, αλλά για το θέμα των... Ε, πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας διατροφικών προϊόντων που αφορούν παχύσαρκα άτομα θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, σε αυτή την νομοθεσία και να μην είναι γενικότερα στα διατηρητικά προϊόντα. Συμφωνεί ε, με τα ε, θέματα της δυσανεξία στη γλουτένη και το πώ θα πρέπει να ρυθμίζονται στον κανονισμό και υποστηρίζει και τι τροπολογίε της εισηγήτριας για τα νανοηλικά. Υποστηρίζει επίση τι διευκρινήσεις τη εισηγήτριας ε, ως προς το ότι κάθε κατηγορία χρειάζεται ε, ένα ξεχωριστό κατάλογο ε, συστατικών. Αλλά όσον αφορά τα βρεμφικά γάλατα και τα γάλατα για μεγαλύτερε ηλικίε παιδιά, εάν έχει αποδειχθεί ότι μία ουσία είναι ευεργετική για την υγεία των παιδιών και έχει λάβει και θετική έγκριση από την ΕΦΣΑ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σε όλους τους ε, σε όλες τις ηλικίε. Αν κάτι είναι καλό για τα βρέφη, θα πρέπει να είναι λογικό να βρίσκεται σε όλα τα ε, προϊόντα αυτής της κατηγορίας και αν κάτι είναι πολύ ακριβό, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορεί να συμπεριληφθεί. Και επίσης θα θέλαμε να περιληφθεί ο κατάλογος αυτός για τα υποχρεωτικά στατικά των βρεφικών τροφών και να περιλαμβάνονται στον υποχρεωτικό κατάλογο. Στη συνέχεια η Τζίλι Γκέρλινγκ ω και εισηγήτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένα τα όσα μα είπε. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε. Έχω ένα-δύο θέματα όμω τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Με ανησυχεί το θέμα της δίαιτας πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας. Αρχικώς είχα την άποψη ότι υπήρχαν ιατρικοί λόγοι και έπρεπε να συμπεριληφθούν αυτά εντός του πλαισίου, αλλά διαρεύνησα πολύ το ζήτημα και αυτό το οποίο ε, έχω κρατήσει είναι ότι όταν προσθέσουμε το κόστος της παχυσυρκίας ε, και όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για καρδιοπάθειες, το διαφύτη και το γεγονός ότι είναι ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα, ε, είδα κάποιες έρευνες οι οποίες κατέδειξαν σαφέστατα ότι τα παχύσαρκα άτομα δεν θέλουν να πηγαίνουν στο γιατρό. Πηγαίνουν 8 ή 9 φορές λιγότερο από ένα άτομο συνήθους βάρους. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ε, ότι είναι λογικό να λέμε ότι θα πρέπει να μπορούν να ε, έχουν δίαιτα πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας ε, και ναι, μεν λέμε ότι έχουν αποτελέσματα για πολύ κόσμο, αλλά όχι για όλου. Ε, δεν είναι λογικό να λέμε ότι θα πρέπει να πηγαίνουν στο γιατρό, διότι όλε οι έρευνε καταδεικνύουν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάνε στο γιατρό, εκτό και αν υπάρχουν άλλε ιατρικέ επιπλοκές. Καλό θα ήταν να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χάσει βάρο πριν φτάσουμε στι ιατρικέ επιπλοκέ. Ε, δεν θα ήθελα λοιπόν να το υποστηρίξω αυτό. Υποστηρίζω την Έστερ για τα θέματα της δυσανεξίας στη γλουτένη και τις βρεφικές ε, τροφές. Ήθελα να σχολιάσω και εγώ τα ίδια πράγματα. Πολλά από αυτά βέβαια αλλάζουν στο νομοθετικό πλαίσιο, τα οποία θα μας οδηγήσουν βέβαια σε λογικά συμπεράσματα στους ισχυρισμούς για τα τρόφιμα, διότι έχουμε πολύ καλό ε, πολύ καλά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση και μετά τα Χριστούγεννα νομίζω ότι θα γίνει και η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπω σε αυτή. Έχω και την ίδια ερώτηση για το θέμα των ε, φυτοφαρμάκων το οποίο ανοίγει ε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο και δεν ξέρω ότι κατά πόσον θα πρέπει να το κάνουμε σε αυτό το κείμενο. Ε, οι καταναλωτές χρειάζονται πληροφορίες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ε, διαθέσιμες πληροφορίες για το κατά πόσον αγοράζουν βιολογικά ή μη προϊόντα και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση εδώ. Ευχαριστώ. Επόμενο ε, σκιώδη ηγητή είμαι εγώ και θα τα πω στα σου ειδικά για να είναι διαφορετικός ο ρόλος μου. Ευχαριστώ την Φρεντερή Κρίση για αυτή τη γνωμοδότηση, όπως και στην πρώτη συνεδρίαση των σκιώδων εισηγητών. Συμφωνήσαμε για τα περισσότερα σημεία και ελπίζω να φτάσουμε σε καλό τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα εδώ να επανέλθω στα όσα είπε η Λίντα Μακάβεν οι κανόνες που έχουμε σήμερα για τα βρέφη, για τα γάλακτα, για τα βρέφη είναι καλά και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να διευρυνθεί για τα παιδιά από 6 έως 12 μήνες. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις για τα τρόφιμα για τα παιδιά αυτά από 6 έως 12 μήνες. Το συζητήσαμε ήδη αυτό. Και νομίζω ότι αυτό θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε ορισμένα προβλήματα αν διευρύναμε αυτήν την ε, ψαλίδα ε, και περιλάβουμε τα παιδιά από 6 έως 12 μήνες. Η επίσης ανέφερε ένα άλλο θέμα. Μίλησε λοιπόν για αυτό που ονομάζεται ε, τα γάλακτα για την ανάπτυξη ε, και νομίζω ότι αυτή η αντίληψη είναι παράλογη. Γιατί να μιλάμε για τέτοια γάλακτα, θα πρέπει να έχουμε μια ειδική κατηγορία και να πούμε περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για γάλακτα αγελάδας με ε, συνθετικές ουσίες που προστίθενται, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω ότι θα μπορούμε να βρούμε μια λύση με βάση τους κανόνες που έχουμε ήδη για όλες τις αλλεργίες και θα πρέπει να προσδιορίσουμε ορισμένα όρια και αυτό που έχουμε σχετικά με την σήμανση να είναι σωστό, ούτως ώστε όσοι έχουν δυσανεξία στη γλουτένη να μην ξεπεράσουν εδώ το όριο των 20 μικρογραμμαρίων ανά ημέρα. για τις δίαιτες μειωμένων θερμίδων, πολύ χαμηλών θερμίδων. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο ε, θα πρέπει όλα αυτά να ρυθμιστούν στο πλαίσιο των, φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών προϊόντων, να υπάρχει μια αναδιατύπωση, διότι εδώ έχετε ορισμένα όρια τα οποία είναι πολύ χαμηλά, θα πρέπει να ξαναδούμε την διατύπωση, διότι εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για ε, μια δίαιτα είναι, η οποία είναι χρονικά περιορισμένη. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος όταν χρησιμοποιείται αυτή η δίαιτα για πάρα πολύ μακρά χρονική περίοδο. Μπορεί να παρουσιαστούν ε, προβλήματα όταν χρησιμοποιεί κανείς πολύ συχνά αυτά τα τρόφιμα ε, ε, είναι, υπάρχει πρόβλημα και η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω στο γεγονός ότι ότι εμένα, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μου ε, βρίσκουν ότι αυτά που αγοράζουν σε κουτιά είναι αειδιαστικά, δεν είναι καθόλου καλά τρόφιμα, είναι κάτι το σημαντικό. Ε, θα περιοριστώ εδώ. Και τώρα, Ανδρέα Σαμονή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεσης και γενικά αλλά και για τη στρατηγική που επέλεξε. Δεν έχω πιστεί όμως απόλυτα στο σημείο στο οποίο ναι μεν εκφράζει ιδιαίτερη ευαισθησία ε, στα άτομα που πάσχουν από κυριοκάκι, ε, δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικέ ανάγκες της ε, συγκεκριμένης αυτής κατηγορίας ασθενών. Από, όπως με επισήμενε ε, η Ιταλική Οργάνωση Πασχόντων από Κιλιοκάκη και πολλοί οργανισμοί ε, και εκπρόσωποι των οργανισμών αυτών, δεν μπορούμε να προσπίσουμε τη λύση που μας ε, παρουσιάζει η συγγήτρια, η οποία ναι μεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά ε, λέει ότι οι κανόνες που αφορούν τη γλουτένη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ισχυρισμό ε, και να βασιστούν στον κανονισμό 1969 του 2011. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει προϊόντα συνήθους χρήσης ε, του υγιούς πληθυσμού και όχι τα προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνουν γλουτένη, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία παράγονται με ειδικό τρόπο για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Όπως είπε και η συνάδελφος Ρης ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα αφορά τις ε, χαμηλής θερμιδικής αξίας δίαιτες, θα πρέπει επειδή ακριβώς υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι διατροφής ε, για συγκεκριμένα προϊόντα, θα πρέπει να διατηρηθούν στην ειδική κατηγορία και τα άτομα τα οποία έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Διότι είναι ένα ε, ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού που ε, πάσχει από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Η κυκλιοκάκη είναι μια χρόνια αναγνωρισμένη ασθένεια και δεν είναι απλώς μια τυχαία δίαιτα. Ο ακαδημαϊκός και ιατρικός κόσμος αναγνωρίζει ότι η διατροφή χωρίς γλουτένη ε, είναι συνταγογραφημένη και καθορίζεται μετά από συγκεκριμένη διάγνωση και μπορεί να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνέπειες εάν κάποιος καταναλώνει γλουτένη να δεν πρέπει και να έχει πολύ σημαντικά εταιρικά προβλήματα ακόμα και ε, με ίχνη γλουτένης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ένα λεπτό έχουμε, θέλουμε να συγκεντρώσουμε την λοιπόν προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου θεωρώ ότι δεν πρέπει να ε, επικαλύπτουμε τα πράγματα. Το ξέρει και ο Καλσλούτερ αυτό. Ότι ε, εξετάσαμε το θέμα του κανονισμού για τα φυτοφάρμακα και ξέρουμε τι υπάρχει εκεί και τώρα έχω ένα πρόβλημα να πούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται εάν υπάρχουν ε, κατάλοιπα τα οποία δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Ε, ναι, αν δεν μπορούμε να τα βρούμε όμως τα κατάλοιπα, τι γίνεται. Και στον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα έχουμε αναφερθεί στις ευαίσθητες ε, ομάδες, ιδιαίτερα τα παιδιά, ιδιαίτερα τις, τις μητέρες, ακόμα και τα γέννητα παιδιά, θα πρέπει νομίζω να το σεβαστούμε και να το αποδεχτούμε αυτό που πετύχαμε με μεγάλο κόπο. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθούμε στους καλούς κανονισμούς που έχουμε ήδη για να τηρήσουμε το ίδιο επίπεδο. Τώρα λέμε ότι τα κατάλοιπα θα πρέπει να είναι λιγότερο από το 0. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν καθόλου ούτε λιπάσματα ούτε φυτοφάρμα. Εγώ έχω πρόβλημα με τα φυσικά, με τα φυσικά δηλητήρια που υπάρχουν. Λοιπόν, σας παρακαλώ να έχουμε το σωστό μέτρο και σταθμό εδώ. Γιατί δεν πρέπει να φτάσουμε στο να μην παράγουμε καθόλου ε, βρεφικές τροφές στην Ευρώπη και να τα εισαγάγουμε όλοι από την Ασία. Λοιπόν, όταν συζητάμε για τα ε, φυτοφάρμακα να το κάνουμε προσεκτικά γιατί έχουμε ένα ειδικό κανονισμό γι' αυτό και έχουμε αναφερθεί εκεί στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καρτίνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, αλλά πρέπει να πω ότι επειδή εμείς οι Ιταλοί, επειδή καταναλώνουμε και πολλά μακαρόνια, πίτσες, ψωμί, ε, προϊόντα δηλαδή που περιλαμβάνουν γλουτένη και είναι βασικά τμήματα της διατροφής μας. Ε, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι ε, για το θέμα αυτό. Τα άτομα τα οποία πάσχουν από κοιλιοκάκι στην Ιταλία είναι πολύ γνωστό. Είναι μια ομάδα που καταναλώνει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Ιταλία και Υπάρχει και πολύ καλή ποιότητα ε, των προϊόντων αυτών ε, από τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας. Όπως υπενθύμησε και ο Ιταλός συνάδελφος, ένα άτομο που πάσχει από κοιλιοκάκι ε, έχει μία διατροφή η οποία αποκλείει πλήρως την ε, γλουτένη μετά από διάγνωση και από ιατρική σύσταση. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να προσπαθούμε να μειώσουμε το επίπεδο ελέγχων για μία τόσο ευάλωτη κατηγορία. Πέρα από τις πολύ ε, σημαντικές ασθένειες τις οποίες μπορεί να πάθουν τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκι αν δεν είναι πολύ αυστηροί στη διατροφή τους, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες συνέπειες, υπογονιμότητα, ε, συνεχής αλοπεκίας, αμβλώσεις, αλοπεκίωση, εγκεφαλικές κακώσεις. Ε, πρόκειται για μια κατηγορία λοιπόν που είναι πολύ εκτεθειμένη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό να καταργηθεί η διαδικασία κοινοποίηση που είναι η μόνη που μπορεί να διασφαλίσει ότι θα γίνεται σαφής έλεγχος για τα προϊόντα. Ο κανονισμός για τους ισχυρισμούς για τη διατροφή δεν το προβλέπει και επομένως θα μειωθεί σημαντικά ο έλεγχος για μια τόσο ευάλωτη κατηγορία. Επιπλέον υπάρχει και μια στρέβλωση την οποία διαπιστώνουμε ήδη. Θα είδατε ίσως κάποιες ε, συνεντεύξεις κάποιων ηθοποιών ε, οι οποίοι λένε ότι από τότε που δεν καταναλώνω ε, γλουτένι νιώθω καλύτερα. Φαίνεται σαν γενικότερο ισχυρισμό που είναι καλός για όλο τον πληθυσμό. Κάτι το οποίο είναι κατάφορο σφάλμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό να μειωθεί το επίπεδο προστασίας όχι μόνο για τα άτομα που πάθουν από κοιλιοκάκι αλλά και για τον όλο πληθυσμό που μπορεί να πιστέψει ότι αν γενικώ δεν καταναλώνουμε γλουτένι είναι καλό για τον οργανισμό κανονισμός μας, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές. Ευχαριστώ. Και πάλι ε, Ιταλός ο επόμενος ε, ομιλητής, ο Ρέστε Ρώση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε η συνάδελφος Γκαρντίνη μόλις τώρα. Μάλλον υποτίμησε το θέμα η συγγήτρια, διότι ε, συνδέει την πρότασή της απλώς και μόνο σε οικονομικά ζητήματα και όχι στην ποιότητα ζωής ανθρώπων που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια. Η κοιλιοκάκη μπορεί να είναι πολύ ε, μικρής επικινδυνότητας, αλλά μπορεί να φτάσει και μέχρι την απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου. Και η συγγήτρια... Ε, θα πρέπει να θυμάται ότι όποιος ζητά να αυτοί που ζητούν συγγνώμη να διατηρηθεί ο κανονισμό για τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκι δεν είναι οι επιχειρήσεις που θα μπορεί να έχουν κάποιο κέρδο ή όφελο, αλλά είναι οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς. Επομένως, οι Ιταλικές οργανώσεις ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκι έχει περίπου το 80% των διαγνωσμένων ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε λοιπόν σε απλά τυχαία στοιχεία, αναφερόμαστε στην μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που μας ζητούν να διασφαλίσουν την πρότητα αυτών των προϊόντων διατηρώντας τα στον κανονισμό. Εάν δεν κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι ασθενείς καταναλωτές, θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και ένα τεράστιο σφάλμα. Ε, η Ιταλική Γερουσία Σα έχω επισυνάψει και το σχετικό έγγραφο, ζητά ακριβώς το ίδιο, διότι ε, στην Ιταλία, όπου τα άτομα που πάσχουν από κοιλιακάκι είναι πάρα πολλά, ίσως πολύ περισσότερα από τις άλλες ε, χώρες μαζί, και τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν πολλά από αυτά τα προϊόντα. Αν εμεί λοιπόν τροποποιήσουμε τον κανονισμό αυτό, ελοχεύει ο κίνδυνο να μην προσφέρονται αυτά τα προϊόντα τα οποία στην Ιταλία θεωρούνται ιατρικά προϊόντα ε, και να μην μπορούν να προσφέρονται πλέον δωρεάν. Επομένω, θα υπάρξει και οικονομική ζημία για του ανθρώπου αυτού, πέρα από ζημία για την υγεία του. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να ξανασκεφτεί αυτό που πρότεινε και να προβλέψει οι καταναλωτέ καταναλωτές αυτοί οι οποίοι μας ζητούν να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων για τα άτομα που πάσχουν από κοιλιακάκι και να παραμείνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαίρετη εργασία, την καλή αυτή βάση συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απλουστεύσουμε και να βελτιώσουμε ε, τους κανονισμούς, αλλά είπε, λέχθηκε και κάτι άλλο. Πρέπει να σκεφτούμε τον τελικό καταναλωτή, τον γονέα που αγοράζει τροφές ε, για το βρέφος ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη σύγχυση για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μην την επιδεινώνουμε. Θα ήθελα να επιμείνω πάνω στο γεγονός ότι πρέπει να απλουστεύσουμε τους κανόνες εμπορίας και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να έχουμε περισσότερη σαφήνια και ίσως να προχωρήσουμε ίσως πολύ περισσότερα από αυτά που προτείνει η συγγήτρια. Να έχουμε ίσως περισσότερη πραγματογνωμοσύνη όταν θέλουμε να δούμε ε, τι ε, γίνεται σε κάθε κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο ε, να βρούμε μια άκρη. Δεν ξέρω ποια είναι τα πλέον Θα πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να πούμε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι προτού δώσω τον λόγο και πάλι ε, για το θέμα των τροφίμων χωρίς γλουτένι, διότι νομίζω ότι το βασικό θέμα στην Ιταλία είναι ότι όταν αναγνωρίζεται ε, ότι ε, είναι έτσι, αυτό υπάρχει επιστροφή για την ασφάλεια. Ε, το θέμα λοιπόν ε, της κάλυψης ε, της επιστροφής, αυτό θα πρέπει να επιληθεί σε ιταλικό επίπεδο. Η ιταλική κυβέρνηση είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν είναι έξω από το πλαίσιο, μπορεί να καλύπτονται. Εμείς δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, η ιταλική κυβέρνηση μπορεί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο είναι αν δεν αλλάξει τίποτα για τον τελικό καταναλωτή, αν τα προϊόντα χωρίς γλουτένη ή με χαμηλή γλουτένη είναι εκτός του ειδικού πλαισίου πλαισίου, στο γενικό πλαίσιο. Τότε έχουμε μια ερώτηση για την Κομισιόν, διότι νομίζω ότι σε πολλά κράτη-μέλη αυτά τα προϊόντα δεν ε, ε, επιτρέπονται, ε, είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές τελικά από, από την γενική νομοθεσία. Να έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήνουμε με το θέμα της κάλυψης στα κράτη-μέλη, δεν ξέρω. Ήθελα βεβαίω να αναφέρω το θέμα αυτό για την Επίτροπη. Είναι μια, ένα ειδικό θέμα της Ιταλίας ε, για την ε, κάλυψη. Είναι κάτι, ένα θέμα που δεν προβλέψαμε, είναι αποτέλεσμα ορισμένων εκστρατιών λόμπι διότι έχουμε πολλά άτομα που είναι, έχουν δυσανεξία στην γλουτένη και στην χώρα μα, αλλά με, την νέα οδηγία για την επισήμανση ε, θα λυθεί το θέμα. Δίνω τον λόγο στην Κομισιόν, αλλά πριν από αυτό ο Κόνη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητή για την πάρα πολύ καλή δουλειά, ποιοτικά. Τα πάντα λέχθηκαν, είχα και εγώ ορισμένε παρατηρήσεις, αλλά έχουν ήδη διατυπωθεί. Αλλά θα ήθελα η Κομισιό να ενθαρρύνει τα κράτη να ασκήσουν κάποια παιδαγωγική στον πληθυσμό διότι έχουμε όλο και πιο πολύ παχύσαρκα παιδιά, το ποσοστό της παχύσαρκίας αυξάνεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τρώνε ε, τηγανιτές πατάτες ε, τα παιδιά, πολλά γλυκά, πίνουν σόδα και οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι ΜΕΣ θα μπορούσαν ε, στην, ε, ε, για τον πληθυσμό που ενέχει κινδύνους να ασκήσουν κάποιο παιδαγωγικό έργο. Θα πρέπει η Κομισιόν να ενθαρρύνει τα κράτη προς το δρόμο αυτό. Το ίδιο πράγμα για την θνησιμότητα στους δρόμους. Η Ευρώπη έχει επίσης μια προσέγγιση παιδαγωγική διδακτική απέναντι στα κράτη ούτως ώστε να μειωθεί το ποσοστό θνησιμότητας στους δρόμους λόγω των τροχέων η Επιτροπή θα μπορεί να το σχολιάσει και αυτό επίσης. Ο κύριος Βασίλης Μαθιουδάκης θα λάβει το λόγο. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με τα θέματα αυτά και υποβάλλετε βάλετε αυτές τις ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Θα ήθελα στην αρχή να συγχαρώ την κυρία Ρίση για τη θαυμάσια περιγραφή του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η πρότασή μας και θα ελπίζω να σας ευχαρώ και εκείνη και τους σκιώδους συζήτητες για την έκθεση που παρουσιάζει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά συνένεση πάνω στις γενικές γραμμές της πρότασης, ιδίως η εξάλληψη της ιδέας των διαιτικών προϊόντων. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρόταση να διατηρηθούν τα τρόφιμα για αδυνάτισμα σε αυτό το πλαίσιο. Ακούσαμε για δίαιτες πολύ χαμηλής θερμιδικής περιεκτικότητας. Ακούσαμε πολλά για αυτού του τύπου τα τρόφιμα γενικότερα. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω ότι η Κομισιόν ακούει προσεκτικά τις ανησυχίες που εκφράζονται. Πιστεύουμε όμως ότι οι ανησυχίες αυτές ε, σχετίζονται με την κατανάλωση αυτών των διαιτητικών προϊόντων αδυνατίσματος που υποκαθιστούν το σύνολο της ε, καθημερινής ε, δίαιτας και όχι κάποια μικρά μικρού τύπου τρόφιμα που τρώγονται διαμέσως, διάμεσα από τα κυρίως γεύματα. Όσον αφορά τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνουν καθόλου βλουτένη, άκουσα τους Ιταλούς ε, βουλευτές που υποστήριξαν την άποψη να συμπεριληφθούν αυτά τα προϊόντα. Θα ήθελα να σας καθησυχάσω συγκεκριμένα εσάς, αλλά γενικά το Κοινοβούλιο, ότι ότι οι κανόνες για εκείνους που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη δεν θα αλλάξουν καθόλου. Ακριβώς οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν σήμερα θα διατηρηθούν με τους ίδιους όρους για, να, την αναγραφή ε, χωρίς γλουτένη ή με πολύ χαμηλό ποσοστό γλουτένης και καλύπτονται αυτοί που έχουν γλυοκάκι νομίζω οι κανόνες και η προστασία για τα άτομα αυτά δεν θα αλλάξει καθόλου. Όπως είπε και η κυρία Λάνε και σήμερα με την ερώτηση σας κύριε Σλότερ δεν επιβάλλουμε καθόλου τη δική μας άποψη στη Βούλη των κρατών μελών για να υποστηρίξουν να υποστηρίξουν οικονομικά την αγορά αυτών των προϊόντων κατά μία τρόπο, όπως ίσως κάποια άλλα κράτη-μέλη αποφασίζουν να επιστρέφουν το κόστος κάποιων άλλων τροφίμων για ειδικές ασθένειες. Εμείς με την πρότασή μας δεν αφορούμε καθόλου τη δυνατότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν να δρουν κατά τον τρόπο που επιθυμούν. Όσον αφορά τώρα τα φυτοφάρμακα, ένα θέμα που εφήγει από όλους σχεδόν τους ε, και την ίδια τη συνεισηγητρία. Θα ήθελα να να αυτό που είπε η κυρία Κλάς. Συμφωνούμε ότι τα φυτοφάρμακα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυτά. Αλλά με το να πούμε ότι απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρμάκων, δεν νομίζω ότι επιτυχάνει το στόχος, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχουν όρια. Αυτά τα όρια του 0,01 ppm που έχουμε σήμερα είναι ένα όριο που υπάρχει στην 396 του 2005 για τα φυτοφάρμακα και είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Γιατί το όριο είναι το όριο ανείχνευσης και έχει εγγραφεί εκεί για να είμαστε σίγουροι ότι φυτοφάρμακα τα οποία ίσως δεν χρησιμοποιήθηκαν αλλά υπάρχουν γιατί υπάρχει μόλυνση των εδαφών από το παρελθόν ή από άλλες ε, καλλιέργειες κλπ. Όλα αυτά ανοιχνεύονται και τα λόγω προϊόντα απορρίπτονται. Αξιότιμα μέλη, μην αφαιρέσετε τη δυνατότητα να υπάρχουν αυτά τα μέγιστα όρια, γιατί αυτά προστατεύουν πολύ καλύτερα από μια διάταξη που θα έλεγε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης, όλοι ανησυχούμε για τις ΜΜΕ. Εάν υπάρχουν κάποιες διατάξεις στα πλαίσια των ισχυρισμών, υπάρχει αρκετή κατεύθυνση Εάν όμως τώρα εμείς υιοθετούσαμε συγκεκριμένες καθημερινές γραμμές με εκτελεστικές πράξεις ή με εντεταλμένες πράξεις όπως κάποιοι νομίζω προτείνουν δεν θα έχουμε κάτι δεσμευτικό και δεν είναι αυτό αυτό που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ. Λοιπόν, ναι, να τις βοηθήσουμε. Να προσπαθήσουμε με νέους κανονισμούς, αλλά όχι με κάτι που θα τους δέσει τα χέρια. Όσον αφορά αυτό το, το μείγμα, ρώτησε κύριε Λάγκα, που είναι για την ανάπτυξη λέγεται και τι θα γίνει να δεν καλύπτεται από τις δικές διατάξεις αυτού του κανονισμού. καλύπτονται βέβαια από του οριζόντιου κανόνε, ισχυρισμοί βάσει των γενικών κανόνων για τα τρόφιμα. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν. Και θα πρέπει φυσικά να υποβάλλεται ένα φάκελος για ένα τέτοιο ισχυρισμό για να αιτιολογείται διακόπτει ο πρόεδρος. Το θέμα του για την ανάπτυξη είναι ισχυρισμός ήδη θεωρείται ναι, μάλιστα. Θεωρούμε ότι κάτι που αναφέρεται στην ανάπτυξη, ανάπτυξη των παιδιών, αναγνωρίζεται μέσα στα πλαίσια του κανονισμού για τους χειρισμούς ότι θα ήταν ισχυρισμός. Καλύπτεται εκεί λοιπόν. αλλά και σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται ε, κάποιοι άλλοι όροι γάλα για παιδάκια ενός με ή κάτι τέτοιο. Πώς θα ε, αποδειχθεί κατά πόσο αυτό το δικό προϊόν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Τώρα αναφέρθηκε το ότι υπάρχει στην αγορά. Υπάρχουν δύο ειδών προϊόντα, από όσο ξέρουμε. Ένα που είναι πολύ κοντά στο γάλα, στο πρώτο ξένο γάλα που δίνεται και έχουν κάποια σύνθεση όσον αφορά τις πρωτεΐνες και άλλα συστατικά που είναι τροποποιημένα από τη ε, το γάλα της Αγελάδας και άλλα που είναι ενισχυμένο γάλα Αγελάδας. Αυτά τα δύο είδη ε, γάλακτος υπάρχουν θα πρέπει λοιπόν κάποιος κανονισμός να έχει τη δυνατότητα να το εξετάσει και να δει πόσο δικαιολογούνται και αιτιολογούνται αυτοί οι ισχυρισμοί. Έκανε η κυρία Μακάβεν κάποιες προ... προτάσεις εξ ονόμου της κυρίας Σάβου θα πρέπει να περιοριστεί η διαφήμιση για το γάλα αυτό και κ. Σλούτερ είπε το ίδιο όσον αφορά τον περιορισμό των διαφημίσεων για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά 6-12 ετών. Έχω να πω ότι αυτά τα θέματα καλύπτονται από το συγκεκριμένο κανονισμό και δεν θα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε σε, αυτό, ε, σε αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού πλαισίου. Και τέλος, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω, ότι οι κανόνες για τους εξαγωγές ορίζονται ξεκάθαρα στα άρθρα 11 και 12 του Γενικής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Αυτά τα δύο άρθρα αναφέρονται στα τρόφιμα και τους σπόρους προσποράς που εξάγονται και τις ζωοτροφές επίσης που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να τηρούνται οι κανόνες εκτός αν η χώρα εισαγωγής έχει διαφορετικές απαιτήσει. Αναφέρεται συγκεκριμένα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες εδώ, ε, μια που υπάρχουν στην νομοθεσία του 2002 για τον νόμο περί των τροφίμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Yes, uh, however... Ευχαριστώ. Βέβαια, εδώ λέει σαφώς ότι αν υπάρχει διάταξη εδώ, προηγείται αυτό που ε, είναι γραμμένο στον κανονισμό. Θα δούμε λοιπόν τι επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Με αυτό να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Ρήφ. παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, στα διάφορα σημεία, αλλά πάρα πολύ εγκατέλειψαν ε, εδώ ε, τη μάχη. Πάρα πολύ σύντομα στην κυρία Ντελόρ αυτό λέχθηκε για τα περιβόητα grown-up milks, τα γάλακτα για την ανάπτυξη των βρεφών. Εγώ διατήρησα το status quo. Δεν νομίζω ότι αυτό αντιποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη ανάγκη θρεπτική, είναι μια, ε, ένας ισχυρισμός υγείας. Ε, υπάρχουν ε, στα διάφορα κρατημέλη πολλές απόψεις. Οι περισσότεροι περιμένουν μια γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ αν είναι θρεπτική ανάγκη, επιχείρημα για μάρκετινγκ. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον αν θέλουν να υπάρχει ένας ισχυρισμός για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει ε, κανένα εμπόδιο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται σε ειδική θρεπτική ανάγκη για ε, την καινοτομία. Θα συνεργαστούμε μαζί, πρέπει να την προωθήσουμε, κυρία Μακάβεν, για τα ε, τρίτα προϊόντα. Απήντησα στην κυρία Ζαρμπού, το είπα στις τροπολογίες 35 και 42 για την διαφήμιση. Απήντησε και η Κομισιόν, κυρία Ζαρμπό, νομίζω στη χώρα τη είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό αυτό. Συμφωνώ αρκετά με τα επιχειρήματά της, αλλά δεν ξέρω αν όλα ε, είναι εδώ η κατάλληλη θέση για να αποκριθούμε σε, ε, σε τέτοια μελήματα. Σχετικά με τους ξεχωριστούς καταλόγους, στις ε, τροπολογίες 50 και 51 απαντάω. Εδώ οι γνώμε ήταν διχασμένες. Αυτή η περιβόητος κατάλογος της ένσης που θα απλουστευτεί, θα ενοποιηθεί και θα είναι πλήρης. Ε, θα πρέπει να προσέξουμε να διατηρήσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά και να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες των πληθυσμών που έχουν εξορισμού ανάγκες διαφορετικές. Σχετικά για τα προϊόντα πολύ ελαττωμένων θερμίδων, εγώ βεβαίως ε, ε, ακούω αυτούς τους παχύσαρκους ασθενείς, το είπα, και εξορισμού για προϊόντα τα, μεταξύ 400 και 800 θερμίδων είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται ένας γιατρικός έλεγχος. Εδώ και πάλι οι πρακτικές στην Ευρώπη διαφέρουν. Σε ορισμένες σούπερ μάρκετ ε, πολλούνται ελεύθερα στην Αμένο Βασίλειο. Στις κατοχώρες η κατάσταση είναι διαφορετική όπως ε, και σε άλλες χώρες. Η ιδέα λοιπόν ε, όπως λέω στην τροπολογία 32 να τα περιλάβουμε στα τρόφιμα για ειδικέ γιατρικές ανάγκες και είναι ένα επιχείρημα που ευσταθεί και υποστηρίζεται από πολλά Προσπαθώ να προχωρήσω γρήγορα, κύριε Σλούτερ, νομίζω ότι συμφωνούσαμε, συμφωνούσαμε σε όλα. Όχι διαφήμιση. Α, εδώ τώρα για το θέμα της γλουτένης για τους Ιταλούς φίλους, μα ο κύριος Ρωσής, Αμονή και η συνάδελφος που δεν είναι πλέον εδώ. Δεν υπάρχει καμία μέλη από πλευράς μας. Έχουμε πλήρη συνείδηση και η Κομισιό επίσης ε, της εκκλήσης της Ιταλίας για το θέμα αυτό, κυρία Λάγκε, επίσης το επισήμενα. Στην Ιταλία καλύπτονται αυτά τα προϊόντα από τις ασφάλειες. Δεν εναπόκειται σε εμά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Το κάνουμε μόνο προτείνοντας, όπως και εγώ, ότι τα προϊόντα αυτά εξαρτώνται από την τροφική επισήμανση και το λέω, υπάρχει μια διαδικασία κοινοποίηση και εξάλλου ο κανονισμός 2009 για αυτό τα τρόφιμα αφορούσε ειδικά δια, ε, διατάξεις σήμανσης. Ε, λοιπόν, είναι κοντά σε έναν κανονισμό, στον κανονισμό που βασίζεται στη σήμανση. Το Γερουσία αναγνώρισε ε, το γεγονός ότι καλύπτεται από την Ιταλική κοινωνική ασφάλιση Νομίζω ότι οι συνάδελφοι του Ιταλικού Κοινοβουλίου πρέπει να κάνουν αυτή την εργασία, ούτω ώστε ω απόρρια τη νομοθεσία μα αυτό το ειδικό προϊόν να καλύπτεται στην Ιταλία και σε άλλε χώρε αν το επιθυμούν. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο των 27 που πρέπει εμεί να λάβουμε αυτό το μέτρο εφόσον προβλέπταν την νομοθεσία μας σχετικά με τα φυτοφάρμακα, συμφωνώ με τα όσα λέχθηκαν, θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί για τον καλύτερο τρόπο και τον μη επαναληπτικό, μη πλεονάζοντα τρόπο, τον πιο φιλόδοξο να ανταποκριθούμε σε αυτήν την φιλοδοξία, γιατί εργαζόμαστε για τον καταναλωτή, όπως λέχθηκε, δεν υπάρχουν όρια, ατελείωτα όρια ή πολύ ελάχιστα όρια φυτοφαρμάκων. Βεβαίως θα πρέπει να απαντήσουμε με αυτόν τον τρόπο στους καταναλωτές. Εμένα μου φαίνεται ότι στην οδηγία 2006 για την οποία ε, έγινε λόγος προβλεπόταν αυτό, υπήρχε σαφής αρχή για τα τρόφιμα, για τα σκευάσματα, για βρέφη κλπ. Ε, νομίζω στην Ετρολογική Σκέψη 18 υπήρχε η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων. Δεν είναι η πρώτη φορά όπως στην αρχή της προφύλαξης που επαναλαμβάνουμε διάφορα πράγματα. Η αρχή της Better Regulation το είδαμε και για τους χυμούς πορτοκαλιών. Ε, επαναλαμβάνω ορισμένα πράγματα. Αυτό δεν είναι ανώφελο. Αλλά πάμε στην ουσία των προτεραιότητων μας που είναι για ε, ευπαθείς πληθυσμού να έχουμε τρόφιμα χωρίς φυτοφάρμακο και την κυρία Εικονή που δεν είναι πλέον και αυτή εδώ. Σημερίζουμε πλήρω, ε, την αποψή τη, Έχουμε εργαστεί για την ε, παχυσαρκία. Είχαμε ε, μια λευκή βίβλο, μια πράσινη βίβλο και εγώ μια έκθεση για την παχυσαρκία και το στυλ ζωής στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια οριζόντια ανησυχία με μέτρα οριζόντια πολλαπλά που αφορούν πολλέ επιτροπέ, αφορούν ορισμένε κοινωνικέ υποθέσει, εκπαίδευση κλπ. Αυτή η ανησυχία είναι παρούσα παντού και εδώ ανταποκρινόμαστε με ένα ειδικό εργαλείο που δεν αποκλεί να ασχοληθούμε και συνολικά με το θέμα και νομίζω ότι τελείωσα. Χαίρομαι που εργαζόμαστε, θα εργαστούμε μαζί για τις τροπολογίες που θα προταθούν, ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Μου φαίνεται αυτό εφικτό. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν οι Δανείοι αυτά. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 18 Ιαρίου για μας, στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 29 Φεβρουαρίου και από εκεί και πέρα θα δούμε, ε, μπορεί να υπάρχει μια θέση στην Ολομέλεια για τις 17 Απριλίου. Ευχαριστώ όλους όσους ε, συμμετείχαν σε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλες τις εκκρεμότητες για την Ιταλία και τη Γλουτένη, να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ όλους όσους λοιπόν αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και τώρα έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα περάσουμε στο σημείο 14 έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εφαρμογές και την, ε, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισμού για ορισμένα φθοριού χαέρια θερμοκηπίου. Θα θυμάστε ότι προσφάτως ε, υπήρξε και ψήφισμα για τις εκπομπές εκτός δοξιδίου του άνθρωπα για να ληφθούν μέτρα πέραν αυτών που έχουμε στον εφιστάμενο κανονισμό και να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και όχι του Κιώτο και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το συζητήσαμε προκαιρού. Ο κύριος Όουεν νομίζω θα μιλήσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Η κυρία Όουεν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα αρχίσω, είμαι από το, την Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα και εγώ, λίγο με Σφάτς. Καταρχήν θα σα ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία αυτή της Κομισιόν να παρουσιάσει την έκθεση για την εφαρμογή επιπτώσει και καταλληλότητα του, του κανονισμού για ορισμένα θεωριούχα αέρια. Ο λεγόμενο κανονισμό ΕΦΚΑΣ. Καθώ επίση να σα παρουσιάσουμε τα τελευταία αποτελέσματα τη συνάντηση του ΕΜΟ 23 του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011 υιοθέτησε η Κομισιόν την έκθεσή της και αξιολόγησε την εφαρμογή της οδηγίας επιπτώσεις και το κατά πόσον είναι κατάλληλη η πολιτική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού F-GAS. Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι αυτός ο κανονισμός που οθετήθηκε το 2006 ήδη συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων Κιώτο. Παρ' αυτά η έκθεση της Κομισιόν τονίζει επίσης ελλείψεις στην εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει αναλάβει δράση εναντί κάποιων κρατών μελών σχετικά. Όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολιτικής ευκάς, η ανάλυση μας καταδεικνύει όταν εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμός αυτός ταυτόχρονα με την οδηγία για τα κινητές μονάδες ε, ε, κλιματισμού θα μπορέσει να βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος του 2050. Ε, και αυτό γιατί αυξάνεται η η δυνατότητα να σταθεροποιηθούν οι εκπομπές ΕΦΚΑ στα σημερινά επίπεδα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αναρωτιέται κατά πόσον η πολιτική ΕΦΚΑΣ είναι επαρκής ε, να εμπνευθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2050. Ο δικός χαρτής για τα χαμηλά επίπεδα άνθρακα καταδεικνύει ότι ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί η μείωση κάτω του 70% σχετικά με τα επίπεδα του 99%. Επίσης, η έκθεση αυτή καταδεικνύει ότι υπάρχουν πολλοί ε, τομείς όπου τα αέρια ΕΦΚΑΣ μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα αέρια που δεν θα έχουν καμία επίπτωση αρνητική στο κλίμα. Γι' αυτό η Κομισιόν θέλει να βελτιώσει τον κανονισμό ΕΦΚΑΣ προβλέπεται αναθεώρηση στο πρόγραμμα εργασία της Κομισιόν για το 2012 και εξετάζεται ε, η δυνατότητα ακολούθησης κάποιας ε, από τις επιλογές μία συζήτηση η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές μας εργασίες. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για την επίτευξη ενό παγκοσμίου ε, ε, μια παγκοσμία συμφωνία μέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Φίλιπ Αόνο που είναι τη ε, της δράσης για το κλίμα για να σας πει τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντηση. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερίσω εν συντομία για την τελευταία συνάντηση για το πρωτόκολλο του Μόντραλ. Έγινε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και κατά βάση κυριάρχησαν οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση για το Ταμείο της Συμφορά των Χωρών Χορηγών που είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία κτλ. Κυριάρχησαν λοιπόν αυτές οι συζητήσεις για τον κατάλληλο προπολογισμό για το 2012-2014. Υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες από τις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν μπόρεσαν να δώσουν και πάρα πολλά οι αναπτυγμένε χώρες λόγω των οικονομικών συνθήκων και μετά από πέντε μέρες διαπραγματεύσεων καταλήξαμε σε ένα ποσό 450 εκατομμυρίων ε, δολαρίων για τα τρία χρόνια, ε, αλλά φυσικά υπήρχαν πολύ έντονες ε, συζητήσεις. Υπήρξε επίσης συζήτηση και για πολλά θέματα πολιτικής, όπως ε, θα θυμάστε ε, οι χώρες της Βορείου Αμερικής και οι χώρες της Μακρονησίας ε, είχαν προτείνει να υπάρχουν κάποια θέματα για τα φθορούχα προϊόντα βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, όπως και τις προηγούμενες χρονιές υπήρξαν αρκετά έντονες συζητήσεις επί του θέματος αυτού. Εξακολουθεί να μην υπάρχει προθυμία από πλευράς αναπτυγμένων χωρών για να συζητηθούν αυτά τα θέματα, ιδίω από την ε, Βραζιλία και την ε, ε, Κίνα, αλλά και από την Ινδία, που είναι κατά τη συζήτηση αυτών των θεμάτων στο πρωτόκολλο του Μόντρελ, για νομικούς αλλά και για άλλους λόγους. Και υπάρχουν και νέες πλευρές, το Q8 για παράδειγμα είναι κατά των συζητήσεων και έχει ταχθεί με αυτή την πτέρυγα. Δεν υπήρξαν λοιπόν επίσημες συζητήσεις ε, για τα ε, φθορούχα αέρια στη συνάντηση του πρωτοκόλλου του Μόντρελ. Υπήρχε όμως και μια μικρή επιτυχία γιατί υπήρξε μια δήλωση την οποία ετοίμασαν ε, οι Ινδονήσιοι που μας φιλοξενούσαν για εναλλακτικέ λύσει, μία δήλωση λύσεις, ε, μία δήλωση που προσπαθεί να κάνει μία μετάβαση προς ε, χαμηλότερης κατανάλωσης ε, τέτοια αέρια και ζητήθηκε να προσυπογράψουν όλοι. Εκατό από τους παρισταμένους την, την υπέγραψαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της υπήρξε και μία απόφαση που έδινε εντολή στο τεχνικό πάνελ και στο πάνελ οικονομικής αξιολόγησης να κάνει μία μελέτη για τις εναλλακτικέ λύσεις ε, για τα φθοριούχα αέρια και συμπεριλαμβάνει και υδροφθοριούχα και υπήρχε αντίσταση και πάλι από πλευράς Βραζιλίας, Κίνας και Ινδίας και τα HFC λοιπόν θα παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη διότι το τεχνικό αυτό πάνελ θα μας ε, κάνει την έκθεσή του του χρόνου. Επιπλέον υπήρξαν και κάποιες άλλες αποφάσεις. Ε, υπήρξε μία απόφαση για τη χρήση μεθυλοβρομιδίους ε, για, για συγκεκριμένους σκοπούς. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συζητήσεων υπήρξε μια απόφαση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πέρασε παρά το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλη αντίθεση από τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία αλλά εδώ ζητάμε περισσότερες πληροφορίες ε, για τη χρήση μεθυλοβρομιδίους μείου για λόγους QPS. Υπήρξαν και κάποιες ε, κλασικές αποφάσεις για τη χρήση του μεθυλοβρομιδίου και όλα αυτά ε, αντιμετώπισαν στεναρία αντίσταση από πλευράς των ΗΠΑ. Ε, καταφέραμε να περιορίσουμε τα ποσά που ζητούσαν αρχικώς. Είδαμε επίσης και ε, χρήση σε συγκεκριμένε βιομηχανίες και σε αντικείμενα τα οποία εισπνέονται και εφαρμογές των συστατικών αυτών και είδαμε και πάλι την αξιολόγηση του τεχνικού και οικονομικού πάνελ και καταφέραμε να εγκρίνουμε τις συστάσεις τους. Τέλος, θα συλλεχθούν στοιχεία και πάλι για τη χρήση των ε, φθοριούχων αερίων σε ε, σκάφη με ξένη σημαία και ότι ορισμένες φορές υπάρχουν εξαγωγές και τι γίνεται με τα λιμάνια και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα με αρκετέ χώρες που έχουν πολλά σκάφη ε, λόγω του συστήματος σημαίας ε, με, που κυκλοφορούν με δική του σημαία αλλά δεν είναι η ιδιοκτησία τους όπως για παράδειγμα τα νησιά της Καραϊβικής ή κάποια νησιά στον Ειρηνικό κενό. σε και γραμμέ λοιπόν ε, κυριάρχησαν κάποια θέματα, υπήρξαν κάποιε χρήσιμε αποφάσει, αλλά δυστυχώ όχι στο βασικό τομέα που μα απασχολεί, το οποίο μα μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Καλέ ειδήσει αυτέ μπορούμε να να, να σταμα... κάνουμε τη μια καμπάνια πριν από τα Χριστούγεννα για να μην αγοράζουμε προϊόντα με μεθυλοβρομίδια. Εάν ε, βεβαίως είναι στην Ευρώπη τα προϊόντα αυτά, δεν έχουν μεθυλοβρομίδιο τα προϊόντα αυτά. Εάν τα αγοράζετε από τις Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να περιλαμβάνουν μεθυλοβρομίδιο. Δεν ξέρω δεν ξέρω αν υπάρχει, είναι παγκόσμια η απαγόρευση ή όχι από το πρωτόκολλο του Μόντραλ. Σχετικά με το μεθυλοβρομίδιο συμφωνήσαμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια μελέτη για να αξιολογήσουμε συνολικά παγκόσμια ε, γιατί χρησιμοποιείται το μεθυλοβρομίδιο, διότι κάτι είναι κάτι που έχει ρυθμιστεί από το πρωτόκολλο του Μόντραλ παρόλο που αυτό έχει ε, ρυθμιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς ε, και σχετικά με κρίσιμες χρήσεις έχουμε εγκρίνει χαμηλότερα όρια για critical use dominations ε, έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε στις φράουλες της Καλιφόρνιας. Αν δεν αγοράσετε λοιπόν φράουλες από την Καλιφόρνια για τα Χριστούγεννα, είσαστε ασφαλείς. Ναι, είπατε ότι οι χώρες ε, της Βορείου Αμερικής έχουν μια πρόταση για βαθμία εξάλληψη και κατάργηση. Ο κύριος Κυλακάκης. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα ε, που το, πολύ λίγα μέλη το συζητούν. Ε, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό διότι έχει μεγάλες επιπτώσεις απάνω στην κλιματική πολιτική και επίσης μας δίνει μια εκτίμηση πολύ ρεαλιστική του τι είναι η πραγματική κλιματική πολιτική ορισμένων αναπτυσσομένων χωρών, κυρίως της Κίνας. Διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η απόφαση να μην συζητηθεί το θέμα δεν είναι επειδή θέλουν να συζητηθεί κάπου αλλού, είναι επειδή δεν θέλουν καθόλου να συζητηθεί το θέμα. Thank you. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις και έχω και εγώ μια ερώτηση. Ξέρετε πότε μπορεί να γίνει μια πρόταση 2012, διότι η Κομισιόν θα κάνει πάρα πολλές προτάσεις το 2012 και θέλω να ξέρω αν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο τώρα, από τώρα. Okay. Um, Πολύ καλά για να απαντήσω στην Λίντα Μακαβάν στην ερώτησή της πρώτα απ' όλα. Ε, τα βορειοαμερικανικά κράτη ετοιμάζονται να ε, προτείνουν μια περίοδο βαθμίας εξάλληψης της Ολομέλειας όπου προσπαθήσαμε να περιλάβουμε το θέμα αυτό στην ατζέντα. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και το, την αρχή ε, της διαδικασίας βαθμίας εξάλληψης. Αυτό έχει καταχωρηθεί σαφώς στις σημειώσεις της συνεδρίασης, στα πρακτικά της συνεδρίασης σχετικά με το να μην υπάρχει καμία συζήτηση. Έχετε δίκιο κύριε Σκυλακάκη, είναι το θέμα πάρα πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα. Είχαμε περισσότερη ευελιξία από τη Βραζιλία και την Κίνα, περισσότερη προθυμία, περισσότερο άνοιγμα για συζήτηση, αλλά η Ινδία είναι πολύ επιφυλακτική, πολύ αρνητική για να συζητηθεί το θέμα και οτιδήποτε έχει ε, σχέση με άνθρακες φθοριούχος. Και ε, βλέπουμε και το Κοβέιτ επίσης που εμπλέκεται σε όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη μάχη. Είναι σημαντικό λοιπόν που έχουμε αυτή τη μελέτη ε, που κατατέθηκε, έγινε δεκτή από τα μέρη και θα παραχθεί του χρόνου και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια βάση για συζήτηση, για να προωθούμε το θέμα, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να απαντήσω στην ερώτηση του Προέδρου και η Λίντα επίση έθεσε πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει κάτι. Ε, είναι στο πρόγραμμα για το 2012, στο πρόγραμμα νομοθατικής εργασίας της Επιτροπής και προβλέπουμε το θέρος του 2012 να υποβάλουμε μια πρόταση. Ευχαριστώ πολύ και είναι το τέλος ε, του τελευταίου σημείου της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, υπάρχει σήμερα μια συνάντηση ανάμεσα στις 3 και την 5 ε, για τις ε, δωρεά, δωρεά ιστών μεταξύ, εδώ σε αυτή την αίθουσα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά θα είναι οι γλώσσες του εργαστηρίου και ε, καλή χρονιά σε όλους. Στις 24 Ιανουαρίου 9 ως 12.30 θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση. Και θα έχουμε μια νέα συντακτική συνάντηση στις 23. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.